Αγαπητοί προσκεκλημένοι και συνάδελφοι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μερικές φορές είμαι ιδιαίτερα περήφανος που προεδρεύω των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και σήμερα είναι μια τέτοια ευκαιρία. Σήμερα τιμούμε τους βραβευμένους για φέτος με το βραβείο Σάχαρο. Είναι μεγάλη, τεράστια τιμή για μας ότι η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να χορηγήσει το βραβείο στον Ολέγκ Κορλόφ, τον Σεργέη Κοβαλιέφ και τη Λουτμίλα Αλεξέγεβα εξ ονόματος της οργάνωσης Memorial και όλων των αγωνιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η απόφαση αυτή η απόφαση αυτή λέγω ελήφθη ομόφωνα. Με το βραβείο αυτό τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τιμούν εκείνους που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα ακόμη αλλά και εκείνους που έχουν χάσει τη ζωή τους στον ίδιο αυτό αγώνα. Την Αταλία Εστεμίροβα που θα έπρεπε να είναι μαζί μας σήμερα όπως και η Άννα Πολιτκόφσκαγια. Οι δολοφόνοι δεν έχουν ακόμη βρεθεί ούτε δικαστή. Κυρίες και κύριοι, στην Ευρώπη ξέρουμε ποια είναι η τιμή της ελευθερίας και της ελεύθερης σκέψης, ελευθερίας της σκέψης. Στις 16 Δεκεμβρίου, 28 χρόνια ακριβώς μετά τις απεργίες στο ρηχείο Βούγιακ όπου δολοφονήθηκαν από τους κομμουνιστές καταλαβαίνουμε ποια είναι η τιμή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πριν από 20 χρόνια στις 16 Δεκεμβρίου στη Ρωμανία άρχισε μια επανάσταση που κόστισε τη ζωή πάνω, σε πάνω από χίλιους ανθρώπους, αγωνιστές της ελευθερίας και αυτούς. Αυτά συνέβησαν σε χώρες που τώρα είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα είναι μαζί μας. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτό το παρελθόν γιατί είναι καθήκον μας να, να προασπίσουμε τις αξίες αυτές. Στην Ευρώπη απολαμβάνουμε την ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία της σκέψης λόγω των θυσιών αυτών. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι, επαναλαμβάνω, μεγάλη τιμή για μένα η χορήγηση αυτή του βραβείου Σάχαροφ στην οργάνωση Memorial. Νιώθω όμως και κάποια πικρία γιατί νομίζω ότι χρειάζονται περισσότερα τέτοια βραβεία στην Ευρώπη. Σήμερα μιλάμε για προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία και γιορτάζουμε και την 20η επέτειο του θανάτου του Ανδρέα Σάχαροφ προς τιμή του οποίου έχει ονομαστεί το βραβείο στη Ρωσία χρειάζονται περισσότερες οργανώσεις σαν το Μεμοριάλ. Ο κύριος Σάχαροφ είχε προβλέψει την πτώση του τείχους του Βερολίνου και τις αλλαγές που θα συνέβαιναν στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Και οι προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία σήμερα ακόμη περιμένουν να κυριαρχήσει η ελευθερία και ο σεβασμός των δικαιωμάτων τους. Αναμένουν περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι χορηγούμε το βραβείο αυτό σε όλους τους Ρώσους πολίτες. Εμείς οι Ευρωπαίοι βουλευτές χορηγούμε κάθε χρόνο αυτό το βραβείο Σάχαροφ για να υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παντού στην Ευρώπη και παντού στον κόσμο. Και εδώ αναφέρομαι στα λόγια του κυρίου Σάχαροφ που είχε πει ότι η ελευθερία του πνεύματος είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό γιατί καταπολεμά τους υποκριτές και τους δημαγωγούς που στηρίζουν ματοβαμμένες δικτατορίες. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε να προασπίζουμε την ελευθερία του πνεύματος και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη. Οι ευρωβουλευτές που έχουν εκλεγεί άμεσα και δημοκρατικά από τους πολίτες των 27 χωρών μελών, εμείς λοιπόν χορηγούμε το βραβείο Σάχαροφ για να υπενθυμίσουμε ότι παντού στον κόσμο αγωνίζονται οι άνθρωποι για να προασπίσουν τις βασικές τους ελευθερίες. Έχει μία αποστολή η Ευρωπαϊκή Ένωση την προάσπιση της ελευθερίας του πνεύματος παντού. Ελπίζουμε η Ρωσία να γίνει εταίρος μας και σε αυτή την προσπάθεια. Και τώρα ζητώ από τον κύριο Κοβαλιόφ να λάβει το λόγο. Ορίστε. Κυρίες και κύριοι, εξ ονόματος της οργάνωσης Memorial θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υψηλή αυτή τιμή που μας περιποιεί με το βραβείο Σάχαροφ. Ως μέλη της Memorial θεωρούμε ότι αυτό το βραβείο απονέμεται όχι μόνο στο δικό μας φορέα, αλλά σε όλη την κοινότητα των αγωνιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία, που τιμάται με αυτό το βραβείο και όλη η ρωσική κοινωνία που υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ και 40 χρόνια παλιά στη Σοβιετική Ένωση και τώρα στη Ρωσία, οι αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν ε, ε, ορθώσει το ανάστημά τους ζητώντας να εξασφαλιστούν οι δημοκρατικές αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν ήταν εύκολο. Τα τελευταία χρόνια έγινε πραγματικά τραγική η κατάστασή τους. Πολλοί έχουν πληρώσει με την ζωή τους τον αγώνα τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απονέμοντας το βραβείο αυτό στην οργάνωση Memorial σκέφτηκε, πιστεύω, κυρίως τους συντρόφους μας, τους φίλους μας που έδωσαν τη ζωή σε αυτόν τον αγώνα. Σε αυτούς αξίζει πιο πολύ από όλους το βραβείο αυτό και το πρώτο όνομα που θέλω να αναφέρω είναι της Νατάλια Εστεμίροβα που ήταν και αυτή μέλος του Memorial η οποία δολοφονήθηκε στην Τσετσενία. Θέλω να αναφέρω το όνομα του κυρίου Μαρκέλοφ και της κυρίας Πολιτόφσκαγια που και αυτοί δολοφονήθηκαν στη Ρωσία ο Νικολάη Γκυρένκο που πυροβολήθηκε στο, στην Αγία Πετρούπολη και ο Μπαμπάβες στο Τουρκεστάν και άλλες προσωπικότητες του κινήματος αυτού θα ήθελα να σας ζητήσω να σηκωθείτε όλοι στην μνήμη των ατόμων αυτών. Ευχαριστώ. Όλοι αυτοί έδωσαν τη ζωή τους ώστε η Ρωσία να γίνει μια πραγματικά ευρωπαϊκή χώρα <clears throat> όπου η δημόσια και η πολιτική ζωή βασίζεται στην ελευθερία έκφρασης όλων των ανθρώπων και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Πέθαναν έτσι και για την Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη χωρίς τη Ρωσία δεν είναι πλήρης. Ελπίζω ότι κατανοείτε ότι όταν μιλώ για τις ευρωπαϊκές αρχές και την ευρωπαϊκή πολιτική κουλτούρα, δεν αναφέρομαι σε αυτή την ορολογία μονάχα με γεωγραφική ή πολιτισμική άποψη και δεν προσυπογράφω μια ευρωκεντρική αντιμετώπιση. Είναι οικουμενικό το σύστημα αξιών το οποίο, για το οποίο αγωνιζόμαστε. Είναι ένα σύστημα το οποίο εφαρμόζεται και για την Ευρώπη και για τη Ρωσία και για την Κίνα και για την Αφρική και όλες τις υπήρους του κόσμου. Η σημερινή στιγμή έχει ένα ιδιαίτερα συμβολικό χαρακτήρα. Το βραβείο αφενός, αλλά και η μέρα κατά την οποία γίνεται η απονομή και η παρουσία αυτών οι οποίοι παίρνουν αυτό το βραβείο καθώς και η προσωπικότητα αυτών που το απένιμαν. Ο Αντρέη Σάχαροφ πέθανε πριν από 20 χρόνια. Ήταν ένας η διακεκριμένος υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σοβιετική Ένωση. Είχε κάνει δύο σημαντικές προτάσεις. Πρώτον, ότι μόνο ξεπερνώντας την πολιτική διχόνοια και αντιπαλότητα θα μπορούσε η ανθρωπότητα να επιβιώσει και να αναπτυχθεί πλήρως θα έχει δυνατότητα έτσι η ανθρωπότητα να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες προκλήσεις και να εξασφαλίσει την παγκόσμιο πρόοδο και ειρήνη. Η δεύτερη πρόταση του Αντρέη Σάχαροφ ήταν ότι η μόνη αξιόπιστη υποστήριξη στις προσπάθειές μας να ξεπεράσουμε τις πολιτικές διαφορές και τις διχόνοιες βασίζεται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυρίως της ελευθερίας έκφρασης, της πνευματικής ελευθερίας. η Ευρωπαϊκή Ένωση, τη οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε την απονομή του βραβείου αυτού όσο ζούσε ακόμα ο Ανδρέη Σαχάροφ, είναι, αν θέλετε, το πλησιέστερο σε ένα έμβριο αυτή της ανθρωπότητας και της διεθνούς κοινότητας που οραματίστηκε ο Ανδρέης Σάχαροφ. Στη Ρωσία έχει γίνει τη μόδας να μιλάμε για ένα ιδιαίτερο ρόλο ιδιαίτερο δρόμο της Ρωσίας, μια ιδιαίτερη πνευματικότητα της Ρωσίας, ακόμα και τις ιδιαίτερες εθνικές αξίες και παραδόσεις. Στον ευρωατλαντικό κόσμο ακούει κανείς πολλές φορές την άποψη ότι η Ρωσία είναι αυτή που είναι εκτός του χώρου των ε, αναπτυγμένων χωρών και ότι θέλει να ακολουθήσει ένα ξεχωριστό δρόμο. Υπάρχουν τέτοιου είδου οικοτολογίε σε σχέση με τη Ρωσία. Αλλά τι πρέπει να πούμε για όλα αυτά. Η Ρωσία, όπω και οι άλλε χώρε του κόσμου, έχει φυσικά το δικό τη δρόμο, έχει τι δικέ επιλογέ για να καθορίσει την παρουσία της στο διεθνές στερέωμα επί τη βάση των παγκοσμίων αρχών. Καμία χώρα στον κόσμο δεν μπορεί να λειτουργεί επί τη βάση αξιών που είναι δανεισμένες από άλλους. Αλλά η σύνδεση της Ρωσίας με την υπόλοιπη Ευρώπη δεν βασίζεται στο ποιος παίρνει ποιες αξίες από ποιον. Θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα αυτό με διαφορετικό τρόπο. Η Ρωσία έχει συμβάλει στον παγκόσμιο πολιτισμό που σιγά σιγά αναδύεται μπροστά στα μάτια μας. Εδώ θέλω να υπενθυμίσω την μοναδική συνεισφορά της Ρωσίας στην πολιτιστική και πνευματική κληρονομιά της Ευρώπης, τον ρόλο που έπαιξαν οι Ρώσοι και μέσα στη Σοβιετική Ένωση για να δημιουργήσουν μια πραγματική κουλτούρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Αντρέη Σάχαροφ τόνισε ιδιαίτερα το ρόλο τη πνευματική ελευθερία και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ανθρώπινη κοινωνία ήδη από το 1968. Και οι ιδέε του πέρασαν σε πραγματικό επίπεδο, σε επίπεδο υλοποίηση από του αντιφρονούντε, από την ομάδα του Ελσίνκη και από τι άλλε ομάδε αγωνιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και η ομάδα του Ελσίνκη εκπροσωπείται εδώ από τη Λουμπμίλα Αλεξέγεβα στα μέσα της δεκαετίας του 1970 αυτές οι οργανώσεις ζήτησαν ανοιχτά να υπάρξει η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι δεν πρέπει να παραμείνει μοναχά κενό γράμμα των διεθνών διακήρυξεων. Προσπάθησαν να, κινητοποιήσουν την κοινή γνώμη και αναγκάστηκε και η εξουσία να δεχθεί ότι έπρεπε να έχουν κάποια ανταπόκριση αυτέ αυτές οι αιτήσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην, Σοβιετική Ένωση. Παραμένουν παρόλα αυτά πάρα πολλά θέματα τα οποία δεν έχουν ακόμα επιληθεί όπως είναι το δόγμα της ανθρωπιστικής επέμβασης και η ανάγκη προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διεθνές επίπεδο. Παρόλα αυτά τα τελευταία 30 χρόνια έχει δημιουργηθεί ένα σημαντικό επίπεδο προόδου που επετεύχθη στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παραμένει πολλής δρόμος όμως να διατρέξουμε. Απλώς θα ήθελα να πω σήμερα ενώπιόν σας ότι κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει τη Ρωσία από τον κατάλογο των Ευρωπαϊκών Εθνών. Η Ρωσία στο τέλος, στο τελευταίο τρίτο του 20ου αιώνα πέρασε σημαντικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τον δημόσιο χώρο, σε ό,τι αφορά τη δημόσια ζωή. Και η δράση του Αντρέη Σαχάροφ δημιούργησε ένα νέο πλαίσιο για το δημόσιο χώρο στη Ρωσία και τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αν σκεφτεί κανεί και την τραγική ιστορία που έχει διατρέξει η Ρωσία στον 20ο αιώνα. Αν ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ήταν η απαρχή τη νέα πολιτική οργάνωση στη Δυτική Ευρώπη που οδήγησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που μέσα σε ένα σύντομο χρονικό ε, διάστημα ξεπέρασε τους κινδύνους της ε, κυριαρχίας των Ναζί. Στην περίπτωση της Ρωσίας η ανάγκη ανασυγκρότησης προσδιορίζεται από τα 70 χρόνια ενός σταλινικού κομμουνιστικού καθεστώτος, ενός καθεστώτος βίας και τρόμου. Υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία της συνειδητοποίησης της κοινή γνώμης στην ε, Ρωσία. Η συνειδητοποίηση για την ανάγκη να υπάρχει ένα πλαίσιο νόμου και η ανάγκη να ξεπεραστεί το σταλινικό παρελθόν στη Ρωσία. Ένα από τα πρώτα κείμενα <clears throat> που δημοσίευσε ο οργανισμός μας ήταν η έκθεση σε σχέση με τη διαδήλωση της 5ης Δεκεμβρίου που έλεγε στο παρελθόν ότι οι έκνομες δράσεις της ε, κυβέρνησης οδήγησαν σε θανάτους Ρώσων και Σοβιετικών πολιτών και τώρα οι πολίτες πρέπει να είναι επάγρυπνοι για όλα αυτά. Αυτή η ιστορική λοιπόν μνήμη που την έχει ενσθενιστεί η κοινότητα των αγωνιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία είναι και εκτιμένο πια και της κοινωνίας των πολιτών σε όλη τη Ρωσία. Νομίζω ότι είναι τεράστια η σημασία τις δράσεις του Αντρέη Σαχάροφ στα τελευταία χρόνια της ζωής του, λόγω και του γεγονότος ότι κατενόησε πλήρως τις ιδιαίτερες πτυχές που έχει η δραστηριότητα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μέσα στη δραστηριότητα του φορέα μας αυτές οι δύο πτυχές της δημόσιας συνειδητοποίησης στη Ρωσία έχουν συγχωνευτεί σε ένα ενιαίο σύνολο. Πιστεύω ότι με την ευκαιρία της 20ης επαιτίου του θανάτου του Ανδρέη Σάχαροφ, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιλέγοντας εμάς ως αποδέκτες του βραβείου Σάχαροφ έχουν δείξει την κατανόησή τους των συγκεκριμένων αυτών στοιχείων της συμβολής του Ανδρέη Σάχαροφ. Θυμάστε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Κομμουνισμό και τον Ολοκληρωτισμό. Το ψήφισμα αυτό όπως και το ψήφισμα του ΟΑΣΕ που ακολούθησε τον επόμενο μήνα σε σχέση με την επανένωση της διχασμένης Ευρώπης κατέδειξε ότι η Ευρώπη κατανοεί απόλυτα ποιο είναι το πνεύμα της εργασίας μας. Εξ ονόματος του Μεμόρια λοιπόν θέλω να σας ευχαριστήσω για την κατανόησή σας. Είναι παράλογη <clears throat> η πολιτική κατάσταση στη σημερινή Ρωσία, όπως καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι το κοινοβούλιο μας, το Ρωσικό Κοινοβούλιο, κοινοβούλιο της χώρας που υπέστη τα πάντινα από την κομμουνιστική στα ελληνική δικτατορία, αντί να υποστηρίξει αυτά τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ΟΑΣΕ, δήλωσε ότι είχαν χαρακτήρα αντιρωσικό. Καταδεικνύει έτσι αυτό το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα ο σταλινισμός δεν είναι μόνο τμήμα του παρελθόντος ένα μεμονωμένο επεισόδιο του 20ου αιώνα για τη Ρωσία. Έχουμε περάσει κάποια χρόνια συγκεχημένης πολιτικής ελευθερίας στη Ρωσία. Αλλά η αντιμετώπιση των ατόμων ως αναλώσιμων που ήταν το βασικό στοιχείο των ολοκληρωτικών καθεστώτων δεν έχει εξαλειφθεί πλήρως. Οι κρατικές αρχές αποφασίζουν χωρίς να σκέφτονται για τις απόψεις των πολιτών στη Ρωσία. Το κατεστημένο είναι μόναχα μια απομίμηση της δημοκρατίας στη Ρωσία έχει όλους τους θεσμούς της ε, σύγχρονης δημοκρατίας, ένα σύνταγμα, πολιτικά κόμματα, εκλογές, διαχωρισμό εξουσιών, ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα, ανεξάρτητη ραδιοτηλεοπτική φορής. Αλλά όλα αυτά είναι μια μορφή απομίμησης, γιατί ένα αντίστοιχο είδος απομίμησης υπήρχε και κάτω από τον σταλινισμό. Δεν πρέπει σήμερα όμως να επαναλάβουμε τα στερεότυπα αυτά της δημόσιας συμπεριφοράς και αντίληψης από την εποχή του σταλινισμού. Εξάλλου τα τελευταία δέκα χρόνια είδαμε όλο και περισσότερο να χρησιμοποιείται η τρομοκρατία. από τις κρατικές αρχές πάνω από 3.000 άτομα έχουν εξαφανιστεί στην περιοχή της Τσετσενίας, έχουν απαχθεί, έχουν βασανιστεί, έχουν εκτελεστεί και έχουν ταφεί ποιος ξέρει πού πολλά από αυτά τα αδικήματα, τα εγκλήματα έχουν γίνει με κεντρική απόφαση και έχουν εκτελεστεί από τις τοπικές δομές ασφαλείας. Πόσοι έχουν τιμωρηθεί για αυτά τα εγκλήματα, ελάχιστοι. Ποιος τους έφερε ενώπιον ενός τακτικού δικαστή. Η Νατάλια Εστεμίροβα και η Άννα Πολιτόφσκαγε ο κύριος Μαρκέλοφ, οι δημοσιογράφοι αυτοί έχουν δολοφονηθεί. Πού βρίσκονται, πού είναι τα πτώματά τους. Είδαμε λοιπόν να υπάρχει όλη αυτή η βία η οποία ασκείται στην Τσετσενία και κινδυνεύει να επεκταθεί και στην σύνολη Ρωσική Ομοσπονδία. Υπάρχουν παρόλα αυτά άτομα λοιπόν τα οποία δεν θέλουν να επανέλθει στο σταλινικό παρελθόν. Αυτή είναι η βάση του αγώνα μας. Πιστεύουμε ότι κανείς δεν μπορεί να ξαναφέρει τη Ρωσία στον δρόμο της ελευθερίας και της δημοκρατίας εκτός από τον ίδιο το λαό της. Είναι ο λαός της, είναι η συνταγματική θεσμή της, είναι η κοινωνία των πολιτών που θα πρέπει να το πράξει αυτό. <clears throat> Και η κατάσταση στη χώρα μας δεν είναι τόσο απλή όσο μπορεί να φαίνεται σε ένα επιφανειακό παρατηρητή. Η κοινωνία μας έχει και τον αγώνα κατά του σταλινισμού και τον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα που είναι πάρα πολύ έντονος. Τι μπορούμε τώρα να περιμένουμε εμεί από την ευρωπαϊκή κοινωνία και την κοινή γνώμη. Ήδη τα διατύπωσε αυτά ο Ανδρέη Σάχαροφ πριν από 20 χρόνια. Είπε ότι η χώρα μου χρειάζεται την υποστήριξή σα αλλά και την άσκηση πίεση. Μια ενωμένη Ευρώπη έχει την ευκαιρία να αντιμετωπίσει με στεναρό αλλά και φιλικό τρόπο τη Ρωσία με υποστήριξη και άσκηση πίεση. Δεν χρησιμοποιεί όμω τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή τη. Να σα δώσω μοναχά δύο παραδείγματα. Καταρχήν, το έργο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο, το, τρόπος με τον οποίο διεκπεραιώνει τις καταγγελίες των Ρώσων πολιτών. Η δυνατότητα προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα έπρεπε να οδηγήσει τα ρωσικά δικαστήρια να λειτουργούν ανεξάρτητα και επί τη βάση γενικών αρχών δικαίου. Αλλά η εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα έπρεπε να είχε άρει τα, τις αιτίες και τα προβλήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πάνω από 100 αποφάσεις έχουν ληφθεί στο Στρασβούργο για τα θέματα αυτά. Και τι γίνεται στη συνέχεια. Η Ρωσία δίνει στα θύματα τις αποζημιώσεις που ζητά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σαν ένα έδος φόρου ατιμορρησίας, αλλά δεν κάνει καμία έρευνα για τα εγκλήματα που έχουν γίνει σε βάρος τους. αυτοί οι οποίοι έχουν κατονομαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τέσσερι στρατηγοί συγκεκριμένα, δεν έχουν τιμωρηθεί, αντίθετα έχουν προαχθεί. Τι άλλο λοιπόν μπορούμε να κάνουμε πέρα από τις χειρονομίες και μόνο του συμβολικού χαρακτήρα. Επίσης πρέπει να σταθούμε και στις σχέσεις της Ρωσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση οι σχέσεις αυτές σήμερα συνοψίζονται στο γεγονός ότι υπάρχει μια διαδικασία διαβούλευσης με τη Ρωσία κάθε 6 μήνες. Έχουμε αξιωματούχους που δεν είναι και στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο που ανταλλάσσουν απόψεις συνήθως μεταξύ, μεταξύ τους αλλά και κλεισμένων των θυρών για θέματα όπως είναι η Τσετσενία, η Λετωνία, η Λιθουανία, η Εσθονία και στη συνέχεια υπάρχει ένα χάσμα για 6 μήνες τόσο και στην Ρωσία όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο οργανώνονται δραστηριότητες των αγωνιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συντάσσουν εκθέσεις και η επίσημη Ευρώπη λέει τι κρίμα που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και παραμένουν σιωπηλοί. Για μένα λοιπόν η απάντηση του τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση της Ρωσίας είναι να δράσει ένα της Ρωσίας όπως θα αντιμετώπιζε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα η οποία έχει δεσμευτεί να τηρήσει μια σειρά υποχρεώσεων και πρέπει να τις τηρήσεις. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση σπάνια αναφέρει συστάσεις εναντί της Ρωσίας για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συνήθω αποσιοποιεί οποιαδήποτε τέτοια σύσταση. Είτε γιατί θεωρούν ότι είναι μάτιο να κάνουν κάτι τέτοιο, είτε επειδή είναι πολύ μεγαλύτερο το δέλεαρ του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Δεν πρέπει όμως η Ευρώπη να παραμείνει σιωπηρή. Θα πρέπει να επαναλάβει και να τονίζει και να επιμένει ότι η Ρωσία θα πρέπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις της. Μπορεί να μην υπάρχει καμία εγγύηση επιτυχίας, αλλά χωρίς αυτές τις προσπάθειες δεν υπάρχει καμιά ελπίδα ότι θα μπορέσουμε κάποτε να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Εάν δεν υπενθυμίζεται όλα αυτά τα θέματα στη Ρωσία, σημαίνει ότι οι ρωσικές αρχές θα θεωρήσουν ότι έχουν πάρει ένα συγχώρο χάρτη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να μην τίθενται τα θέματα αυτά στην ημερήσια διάταξη της Ευρώπης, αυτά θίγουν την Ρωσία, αλλά θίγουν εξάλλου εξίσου και την Ευρώπη γιατί υπονομεύουν τη δέσμευση των ευρωπαϊκών θεσμών στις ευρωπαϊκές αξίες. Το βραβείο το οποίο απονείμαται σήμερα είναι το βραβείο για την ελευθερία της σκέψης. Πώς μπορεί κανείς να μην είναι ελεύθερος σε ό,τι αφορά τη σκέψη του. Ποιος μπορεί να περιορίσει την ελευθερία σκέψη και πώς. Αλλά παρόλα αυτά γίνεται πολλές φορές γιατί είναι ο φόβος ο οποίος από... γίνεται κάποια στιγμή ένα τμήμα της ανθρώπινης προσωπικότητας και λογοκρίνει, αυτό λογοκρίνει και την ίδια την ανθρώπινη σκέψη. Πολλοί φοβούνται, πολλοί όπως ε, είπε και ο Τζορτζ Όρουελ στο 1984, τελικά κύπτουν την κεφαλή ενώπιον του μεγάλου αδελφού, του Big Brother. Αυτό είδαμε στο σαλινισμό, στον ναζισμό, αυτό βλέπουμε και στην περίπτωση της Τσετσενίας που έχει οδηγήσει στην εξάπλωση ενός κλίματος φόβου σε όλη την Ρωσία. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το φόβο. Μόνο με την ελευθερία της σκέψης. Αυτή ήταν η προσέγγιση του Αντρέη Σάχαροφ. Έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το φόβο. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ελευθερώσουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους από το φόβο. Η ελευθερία σκέψης είναι το υπόβαθρο όλων των ελευθεριών. Γι' αυτό είναι πρέπον το βραβείο Σάχαροφ να είναι το βραβείο της ελευθερίας σκέψης και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που μας το απονείματε σήμερα. Ευχαριστώ. спасибо. Желаем успеха. И вы сделали многое для нас. Ну, Мы да. вам очень благодарны да. и желаем успеха тоже. I would like to congratulate you as well. It was all these people which are awarding uh, awards to you, madam. Thank you.